τα πρακτικά της ε, χθεσινής ε, συνεδρίασης ε, και τα κείμενα που εγκρίθηκαν είναι στη διάθεσή σας. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο σχόλιο από αυτόν.